El señor presidente. Buenos días, amigas y amigos, colegas. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως και ως πρώτο σημείο προβλέπεται η έκθεση του κυρίου Κάλφιν για τη χορήγηση εγγύησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσουμε χθες μέσα το λόγο στον κύριο Κάλφιν. Κύριε Κάλφιν, γνωρίζετε πως έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας προβλέπονταν έξι, αλλά δύο θα σα δοθούν στο κλείσιμο τη συζήτηση. Τώρα, εάν θέλετε να μιλήσετε έξι λεπτά τώρα στην εισαγωγή, εντάξει, δεν θα έχετε στο τέλο χρόνο να μιλήσετε. Για άλλου, τέσσερα συν δύο στο τέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η παρούσα εντολή τη Ευρωπαϊκή Τάξη Απενδύσεων για τι επιχειρήσει εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω εκπνέει τέλο Οκτωβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν επί των συνθήκων και των όρων για την παράταση τη της ε, εντολή πέραν αυτή τη ημερομηνία. Συνήθισε διεξοδικά το Κοινοβούλιο επί σειρά μηνών το θέμα. Κατά τη διάρκεια αυτή συζητήσαμε πάρα πολλέ ιδέε και προσπαθήσαμε να ακούσουμε τι απόψει πολλών εμπλεκομένων μερών. Είχαμε πάρα πολλέ συναντήσει και εντό και εκτό του Κοινοβουλίου ε, οι πολιτικές ομάδες συναντήθηκαν και επεξεργαστήκαν το κείμενο. Εδώ είναι ο χώρος, ε, το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων και από τη διοίκηση για την αφοσίωσή τους και το ότι εργάστηκαν σε πολύ υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και κατέβαναν προσπάθειες να πετύχουν μεγάλη ε, γενικότερη συνένεση όσον αφορά την εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να κάνει τελικά τη διαφορά όσον αφορά την επιτυχία του στόχου της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για την υποστήριξή τους και τις συμβουλές τους που ήταν πολύτιμες για το έργο μας. Τώρα έχουμε ένα σχέδιο αποφάσεω που πρέπει να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο που προβλέπει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και των άλλων φορέων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, καλύτερη ε, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, απόφαση που θα βελτιώσει την ορατότητα των αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων τη Τραπέζη. Με αυτή την απόφαση θα ξεκινήσουμε την επεξεργασία κοινή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με το Συμβούλιο. Το σχέδιο αποφάσεω προβάλλει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων θεωρείται σαν τράπεζα επενδυτική και διεθνής χρηματοστικός οργανισμός. Είναι νέος θεσμός όμως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται να συμβάλλει με καλύτερο τρόπο για την επίτευξη στόχων της ενώσεως με τα εργαλεία που διαθέτει και τα μέσα της. Οι αλλαγές που προτείνονται βασίζονται στη σωρευμένη εμπειρία και την κατανόηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που επενδυτική τράπεζα, δεν θα πρέπει να υπονομευθεί ως θεσμός προτείνει καλύτερο συντονισμό το Κοινοβούλιο μεταξύ τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Τραπέζη αντί εφαρμογή τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώση και των στόχων αυτή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να, να αναπτύξει παραμέτρου ανάπτυξη ε, και επίτευξη στόχων και θα συμβάλλει έμεσα στην εκρίζωση της φτώχειας και την μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος σε αναπτυσσόμενες χώρες και να τονώσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων. Το σύστημα ελέγχου και εποπτείας εγγυάται μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και αυξανόμενες δυνατότητες για τις εμπλοκόμενους φορείς να γνωμοδοτούν σε αρχικό στάδιο τη εξέταση των προγραμμάτων και των σχεδίων άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τα διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Θα πρέπει να συμβάλλουν τα χρήματα αυτά στην, στην προσπάθεια των εταίρων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε προσπάθειε να εφαρμόσουν πολιτικέ που έχουν με το κλίμα. Α ελπίσουμε ότι αυτό το νέο μέσο θα δημιουργήσει κίνητρα για τι χώρε αποδέκτε, ούτω ώστε να, αντι... να προσπαθήσουν να πετύχουν περισσότερου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το κλίμα. Προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση μια αύξηση των ατοτορίων των εγγύσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που θα χρησιμοποιεί η Τράπεζα σε μια πρώτη ματιά αυτό είναι πολύ δύσκολη απόφαση διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για τα κράτη-μέλη μια αύξηση των ατότων ορίων σημαίνει 9% συμμετοχή στο Ταμείο Εγγύσεων. Από την άλλη πλευρά, αυτή, αυτό είναι ένα άριστο μέσο που δημιουργεί φαινόμενο μόχλευση και θα μπορέσουν περισσότερα επενδυτικά ιδρύματα να συμμετέχουν στις προσπάθειε. Η αύξηση είναι περίπου 1,7 δι, η αύξηση τη οροφή, και έτσι η τράπεζα τουλάχιστον θα μπορέσει να διατηρήσει την ένταση των δραστηριοτήτων στι προενταξιακές χώρε και κυρίω στην περιοχή τη Μεσογείου. Τα τελευταία χρόνια, κατόπιν τύπο του Συμβουλίου, η χρηματοδότηση είχε εντατικοποιηθεί. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει και άλλε προσπάθειε για να υποστηρίξει τι προσπάθειε των χωρών των Δυτικών Βολκανίων και τη Βορείου Αφρική, κυρίω του καιρού που περνάμε. Αυτό δεν συνεπάγεται σημαντικέ δαπάνε, ενώ τα ωφέλη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε αυτέ τι χώρε θα είναι πολύ μεγάλα. Ζητούμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δημιουργήσει δυναμικό για την αξιολόγηση και ενημέρωση όσον αφορά την ανάπτυξη, των περιβάλλων και τι πτυχέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά τα προγράμματα που εφαρμόζουν. Θα πρέπει εκείνοι που δανειοδοτούν να συζητούν με του τοπικού φορεί πριν αναπτύσσουν τα προγράμματα και τα προτείνουν. Είναι καλό να μην συνεργάζεται ε, με εταίρους ε, που κινούνται ε, σε φορολογικούς παραδείσους και δεν είναι σαφείς οι όροι τους οποίους κινούνται. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό των πόρων των διαφόρων διανεκδοτών μέχρι τα μέσα του 2012. Θα δημιουργηθεί ομάδα εργασία που θα το αναλύσει αυτό και θα προσπαθήσει έτσι να αυξήσει την αποδοτικότητα των προσπαθειών τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως. όσον αφορά την παροχή βοηθεία σε όλο τον κόσμο. Ε, Το λόγο έχει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ο αντιπρόεδρος αυτής, ε, κύριος Κάλλας. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κάλφιν, αλλά και τα άλλα μέρη του Κοινοβουλίου για την επικοδομητική προσέγγιση της εκθέσεως αυτή που, αυτής που τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη η έκθεση προκειμένου να προχωρήσουμε στι περαιτέρω διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Τον περασμένο Απρίλιο η Κομισιόν εξέδωσε ε, μια τροπημένη πρόταση για την τροποποίηση της πρότασης 23 2009 μετά από ενδιάμεση αναθεώρηση της εξωτερικής εντολής της ε, ΕΤΕΠ. Χρειάζεται λοιπόν να λαμβάνονται αγκαίρως αποφάσεις προκειμένου η ΕΤΕΠ να προχωρήσει τις εξωτερικές δραστηριότητε της μέχρι το 2013 και να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα της κλιματολογικής αλλαγής και της ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σημερινή ψηφοφορία, ε, πολλές ε, τροπολογίες ε, γίνονται δεκτές από την Κομισιόν, τροπολογίες που αφορούν στον ενίσχυση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ δεύτερον να υπάρχει ανάπτυξη των ανωτάτων ορίων αυτό θα οδηγήσει στην, επιτρέψει μάλλον στην ΕΤΕΠ να προχωρηθήσει διάφορε δραστηριότητε ιδιαίτερα στον τομέα των προενταξιακών. Επίσης θα βοηθήσει την ΕΤΕΠ να λάβει μέρο στην κοινή μα προσπάθεια για να παρέχει βοήθεια στην την Ισία και την Αίγυπτο στην διαδικασία εκδημοκρατισμού. Επίση, απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι υπόλοιπε τροπολογίε θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσει στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου. Αυτά τα σημεία άπτονται αφενό στον περιορισμό τη επιλεξιμότητα σύμφωνα με την εντολή για τι κλιματολογικέ αλλαγές από κράτη τα οποία δεν έχουν δεσμευθεί ακόμα για την επιτεύξη κυβέρνων στόχων. Ε, τα τροπολογίε που αφορούν τι περιφερειακέ κρατικέ γραμμέ ω πράξη κατεξιοδότηση που δεν μπορούν να είναι επιχειρησιακές όπως αρχικά είχε προβλεφθεί από την πρόταση της Κομισιόν και τρίτον ορισμένες τροπολογίες που άπτονται ε, θεμάτων μακροπρόθεσμων όπως η δημιουργία μιας πλατφόρμας για περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη αλλά και τις αντανακλάσεις της ε, ε μακροπρόθεσμες δύο προβλέψεις Αυτά δεν αφορούν την ε, ισχύουσα εντολή. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί, διότι αυτέ οι τροπολογίε θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την λήψη απόφαση και θα μα οδηγήσουν σε ε, χρονοβόρε διαπραγματεύσει. Ο τριμερή διάλογο ανάμεσα στα θεσμικά όργανα θα ξεκινήσει με βάση την έκθεση που θα εγκριθεί σήμερα και κοινό στόχο είναι να υιοθετηθεί η απόφαση πριν από το, τέλος, το έτσι ώστε να μπορέσουμε να χωρίσουμε από τον Οκτώβριο 2011 χωρίς να διακόψουμε τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ σε αυτά τα κράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμο μέλη. Ευχαριστώ Επίτροπο, μάλιστα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για δύο ε, λεπτά και τρία δευτερόλεπτα ο κύριο Πεγιό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον συνάδελφό μου τον κύριο Κάλφιν για την έξοχη δουλειά που κάναμε μαζί και εν ονόματι τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας υπήρξα συγγητής του συναδέλφους κυρία Οτάλα, τον κύριο Λάμσντορφ και την κυρία Γιαννάκου. Δεν θέλω να αναφερθώ εκ νέου στα θετικά στοιχεία τη εκθέσεω και τη προτάσεω που υπερασπίστηκε ο κ. Καλφίν. Την συνέταξε ο ίδιο για την εντολή αλλαγή του κλίματο, την αύξηση των ανθρωπίνων πόρων την προσοχή πρέπει να δοθεί στην ε, ανάπτυξη, κοινωνικές, περιβαλλοντικές πτυχές, ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εγγύησει θα πρέπει να επικοινωθούν επί των χωρών που χρειάζονται περισσότερε ανάγκε και χρειάζεται καλύτερη διάθρωση με τι πολιτικέ τη ενώσεω. Πάνω αυτά τα σημεία το είναι ενωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να παραμείνει ενωμένο στι δύσκολε διαπραγματεύσει που αναμένονται έναντι του Συμβουλίου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα επί δύο κενών που υπάρχουν, ανεπαρκείων μάλλον σε αυτή τη φάση. Λυπούμε που τις ψήφισε στη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δηλαδή την ανάγκη ήδη να ετοιμαστεί για μικροπιστώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεν συμπεριελήφθη αυτό το στοιχείο και την ανάγκη ήδη να ξεκινήσουν συζητήσει επί του ανώτατου ορίου μετά το 2013 και γι' αυτό η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών απεφάσισε με τη συμφωνία του συγητού του κ. Κάλφιν και των άλλων εισηγητών να καταθέσει τροπολογίε στην Ολομέλεια επί των δύο θεμάτων. Τέλος υπάρχει κάτι κρίσιμο επί το οποίο θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή, είναι πολιτικής φύσεω και συζητείται επί σειρά ετών όταν το τείχο του Βερολίνου κατέρευσε αντιδράσαμε και με το πρόγραμμα της διευρύνσεως που συζητήθηκε λεπτομερώς και που χρειαζόταν να γίνει αλλά δημιουργήσαμε την BERD ε, για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση που χρειαζόταν, την οικονομική και την πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν πρώτη ε, που έδωσε δάνεια και στην άλλη πλευρά του, της Μεσογείου. αυτή οι πόροι και αυτά τα ταμεία δεν ξεπερνούν ε, μια, ένα προγραμματισμό μέχρι το 2013 και η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα δείχνει ότι ίσως αύριο να υπάρξουν δυσκολίες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη και για την Ένωση για τη Μεσόγειο που συζητείται σήμερα και αφορά και την έκθεση Κάλφιν και αφορά τη δημιουργία μιας ευρωμεσογειακής τραπέζος συν και επενδύσεων είναι ρεαλιστική προσεγγίση πέρα των ρητορικών σχημάτων, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύσει το μεγάλο δημοκρατικό κίνημα που ε, παρατηρείται στην άλλη πλευρά τη Μεσογείου και θα ήθελα κάτι να κάνουμε ε, ούτω ώστε πραγματικά να υλοποιηθεί αυτή η τράπεζα στου επόμενου μήνες. Ευχαριστώ, Βενσόν, για δυόμιση λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριο Μπέρμαν Τάι, Επιτροπή Ανάπτυξη. Πρόεδρε, η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, δεν αγγίζει πολλές ε, ομάδες ανθρώπων και στην Αφρική που είναι, διπλάς, είναι ε, διψήφιος ο ανάπτυξης υπάρχει μεγάλη αύξηση τη ανισότητα, γιατί οι γυναίκες και οι αγρότες δεν έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν τη ζωή τους. Ένα από τα μεγάλα εμπόδια είναι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες γιατί οι ιδιωτικέ ε, τράπεζες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους επιχειρήσεις παρά στις γυναίκες και στους αγρότες. Και εδώ είναι σημαντική η ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η τράπεζα δεν είναι μόνο συνώνυμα των φραγμάτων, των μεγάλων project υποδομής θα πρέπει να συνεχίσουν αυτέ οι δραστηριότητε στι τράπεζε, αλλά φυσικά θα πρέπει να ακούγονται και όλοι οι τοπικοί φορεί και να ακολουθούν τα κριτήρια τη κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα. Δεν ήταν το να επιτρέπουμε φορολογικού παραδείσους. Η ΕΤΕΠ λέει ότι θα ταχθεί υπέρ των πολιτών και μικρών project προκειμένου να του ανοίξει την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των τοπικών τραπεζών μέσω των ε, μικροπιστώσεων και μέσω ε, συνεργασίας ανάπτυξης με αναπτυξιακές τράπεζες. Ε, η ΕΤΕΠ θα πρέπει να έχει το απαραίτητο προσωπικό και την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αλλά η ΕΤΕΠ θα πρέπει να αποτελεί και ένα εργαλείο εκ των άνευ σε αυτή την καινούρια της διάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες για να πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ την ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ και όλους τους συζητητές για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπέρμαν. Από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ένα λεπτό, ο κύριος William Dartmouth. Πρόεδρε, μέχρι τώρα οι επαγγελματίες οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, λειτουργούσαν την τράπεζα με μια κουλτούρα χρηματοπιστωτικής ευφροσύνης. Ε, δινόταν ε, δάνεια και πιστώσεις μεσόφρονα τρόπο και γι' αυτό ήταν λίγα τα κακά δάνεια τα οποία είχαν σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωστόσο αυτό που θέλει να κάνει η έκθεση είναι να αποδυνομήσει αυτή την επαγγελματική κουλτούρα της ΕΤΕΠ και να διευρύνει την εντολή της για να περιλαμβάνει ένα, μια σειρά πολιτικών στόχων. Η χαλάρωση αυτής της ε, εμπορικής ε, κουλτούρας βάσει της οποίας λειτουργούσε ως τώρα η τράπεζα, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε έλλειψη τέτοιων εγγύησεων και αυτό θα κοστίσει στον φορολογούμενο και θα πρέπει εκ νέου να αναρωτηθώ καθώς πόσο οι φορολογούμενοι της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματικά θέλουν τα χρήματά τους να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη πολιτικών και μόνο στόχων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δεν βλέπω στο έδρανό του τον συνάδελφο Τάμα Ντόιτς που πρόκειται να μιλήσει εξ όνομα τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Θα δώσουμε το λόγο για ένα λεπτό τον κύριο Κούτας θα μιλήσει εξ όνομα τη Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέσω της εγγύησης που προσφέρεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεχίζουμε την ε, ανάπτυξη των υποδομών αυτής αλλά και τη μείωση των βελτίωση μάλλον των δομών και υποδομών στα τρίτα κράτη τρίτα κράτη-μέλη αλλά και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι η παράταση της εντολής προς την τράπεζα είναι κάτι το θετικό αρκεί να συμπεριλαμβάνονται τα, οι χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο αλλά και κράτη τα οποία έχουν συνάψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ανάγκη από περισσότερα κονδύλια και από εξειδικευμένα στελέχη και προσωπικό. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη την σημασία που έχουν στρατηγικά σχέδια όπως ο αγωγός ε, Ναμπούκο κλπ πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι η τράπεζα χρειάζεται να παρακολουθεί και να υποπτεύει την εξέλιξη των προγραμμάτων αυτών αλλά και την διαχείρισή τους. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Ντόιτς δεν έχει έρθει ανάμεσά μας. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές που θέλαμε το λέω ξανά των πολιτικών ομάδων. Πρώτος αγορητής, ο κύριος Κολίνο, έχει δύο λεπτά για να μιλήσει στο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κάλφιν, για την εργασία του. Με τη σημερινή ψήφο ανανεώνεται η ε, ε, κοινοτική εγγύηση στην ε, την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύηση για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αποκτά η μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή οικονομική συγκυρία, διότι υπάρχουν βαθιές αλλαγέ όχι μόνο στι αγορέ, αλλά και στην λογική παραγωγή και τον τρόπο σκέψης, τρόπο αντίληψη τη οικονομία. Εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, έχει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει περαιτέρω αυτών των ε, αυτής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση που διεξήχθη ήταν όντω επικοδομητικά τόσο ε, στο πλαίσιο της Τροπής Προπολογισμών όσο και εν ώψη τη προπαρασκευαστικής εργασίας της σημερινή συζήτηση. Η πολιτική άλλη παράθεση αφορούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ε, βελτιστοποίηση των συνεργειών στο πλαίσιο της ε, ανάπτυξης και ώστε παρεμβάσεις να μην ε, επικαλούνται και να μην επικαλύπτονται και να μην υπάρχει σπατάλη πόρων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει δάνεια και ανταγωνίζεται σε διεθνές αγορές και δεν ε, δίνει, κάνει δωρές οι δραστηριότητε λοιπόν της ΕΤΕΠ που έχουν επεκταθεί σε χώρες όπως την Λιβύη και το Ιράκ αλλά όχι σε χώρες όπως η Λευκορωσία ε, που όπου η τήρηση και σεβασμός των τοπικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση. Υπάρχει κάθε ενδιαφέρον και συμφέρον να ε, μπορέσουμε να πετύχουμε την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο των ε, εργασιών ο εισηγητής θα υποβάλει μια προφορική ε, τροπολογία για τις δραστηριότητε της ΜΠΕ και την κάλυψη των ζημιών από χώρες, στις χώρες μάλλον της Μεσογείου και αυτό εν ώψη των ε, προβλημάτων της ε, τελευταίας, ε, των τελευταίων εβδομάδων εν ώψη των μεταναστευτικών ρημάτων. Νομίζω πως ο κύριο Ντάρμουθ επιθυμεί να κάνει μια ερώτηση σχετικά με την γαλάζια βίβλο. Κύριε Ντάρμουθ, παρακαλώ. yes, sir. Um, does the... Ναι, ο αγορητής θέλει να εξετάσει ποιο είναι το κόστος όλων αυτών για το φορολογούμενο. Ε, Μπορείτε να απαντήσετε. Τι θέλετε να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή γενικά. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαντήθηκε ε, ερώτηση και το λόγο τώρα έχει ο επόμενος αγορητής, ο κύριος ε, Φάρμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Κάλβιν. Έκανε έξοχη δουλειά. Εργάστηκε πάνω στο θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συνεργάστηκε με τους κοιόδη εισηγητές του Κοινοβουλίου και με την Τράπεζα. Έκανε έξοχη δουλειά. Η χρηματοπιστική κρίση κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς σταθερούς δημόσιους θεσμούς που παρέχουν πιστώσεις για σημαντικές επενδύσεις όταν η ιδιωτική αγορά είναι ασταθής αναφερόμαστε συχνά στη δημιουργία νέων χρηματοστηρικών μέσων και την εξέλιξη αυτών που διαθέτουμε. Εδώ αναφερόμαστε στη ρίο της Ευρωπαϊκή Τάπεζας Επενδύσεων εκτός Ευρώπης. Να τονίσω κάποια σημεία που ελπίζω να εισακουστούν και εντός Κοινοβουλίου και εντός Συμβουλίου. Καταρχά, αυξημένη συνεργασία μεταξύ δραστηριοτήτων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και των κατευθυντήριων γραμμών για την αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεύτερον, αύξηση του, της οροφής για προγράμματα που αφορούν το κλίμα και τρίτον χρειαζόμαστε αύξηση των εγγύσεων που καταβάλουν τα κράτη-μέλη. Το μεγαλύτερο μερίο της δουλειάς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι στην Ευρώπη. Αν δείτε όμως τον αριθμό χωρών που δέχονται τα δάνεια, οι περισσότερες είναι αναπτυσσόμενες χώρες και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αυξήσουμε τα πρότυπά μας όσον αφορά την αξιολόγηση των προγραμμάτων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αξιολογεί καταρχάς πριν χορηγηθεί η πίστοση κατά πόσο η επένδυση πληρεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει να αυξηθεί επίσης η διαφάνεια όσον αφορά στη θηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όσον αφορά την εντολή για εξωτερική δράση. Για την ώρα έχουμε πολύ περίπλοκες συναλλαγές οικονομικές, οπότε είναι δύσκολο να επικρατεί η διαφάνεια. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά ε, του φορολογικού παραδείσου. Να υπάρχει ευαισθητοποίηση των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα καλό χρηματοδοτικό ε, σύστημα είναι προαπαιτούμενο για εύρυθμη λειτουργία των οικονομιών στον κόσμο και γι' αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε και τι προφορικέ τροπολογίε τι σχετικέ που ελπίζουμε να τι υποστηρίξουν όλοι, οι οποίε τροπολογίε θα μα επιτρέψουν να διαθέσουμε περισσότερου πόρου σε χώρε όπω είναι η Αίγυπτο και την Ισία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στη κατεύθυνση και ελπίζω το Συμβούλιο να το υποστηρίξει στι επικείμενε διαπραγματεύσει. Ευχα... Ευχαριστώ. Εξ των φιλελευθέρων για δύο, δύο μισή λεπτά το λόγο ο κύριος ε, Χαρτμούντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έκανε έξοχη επαγγελματική δουλειά πάνω σε αυτή την έκθεση. Συνεργαστήκαμε όλες οι ομάδες και το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Ακούσαμε διάφορες απόψεις στην αίθουσα. Κάποιοι εξέφρασαν ανησυχίες όσον αφορά ενδεχόμενο υπονόμευση του καλού έργου που επετέλεσε η, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά το παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι είναι αβάσιμε οι ανησυχίε που εκφράστηκαν. Νομίζω ότι κινούμαστε στην ισχύουσα εντολή που έχει δοθεί και θα κατευθύνουμε στο μέλλον την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προ ε, καλύτερου προσανατολισμού. Εκφράστηκαν πολλέ καλέ ιδέε και είναι καλό να θυμόμαστε ότι χρειάζεται να διαπραγματευτούμε την εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύων για το 2014 και πέρα, για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό είναι το υπόβαθρο βάσει του οποίου θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα καθήκοντα και τις εντολές που θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της επομένης χρηματοστικής περίοδου και ποιους πόρους θα απαιτήσει αυτή η τράπεζα. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν στο παρόν πλαίσιο να αναφερθώ σε κάποιες λεπτομέρειες Τη μία την ανέφερε ο κύριο Φέρν. Δηλαδή ότι ίσω θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί αυξήσεως των πόρων, ούτω ώστε η τράπεζα να μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρου αυτού στη Βόρεια Αφρική. Πολύ καλή ιδέα αυτή και κάτι τέτοιο δικαιολογεί και την εξωτερική εντολή που χορηγείται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα να τονίσω επίση και κάτι που ο συνάδελφο μου, ο κύριο Λάμσντορφ, θα πει πιθανότατα σύντομα, δηλαδή ότι η ομάδα των φιλελευθέρων δεν θέλει να χρησιμοποιεί τους πόρους της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δανείσει χρήματα στη Λευκορωσία. Συνάδει και με τις αρχές που υποστηρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η προσέγγιση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και πρέπει να σέβεται κάποιες αρχές. Συνοψίζοντα, πρέπει να πω ότι συνεργαστήκαμε άριστα οι διάφορε πολιτικέ ομάδε, έκανε έξοχη δουλειά ο συγητή, βρήκε πολύ σημαντικέ λύσει που θα μα επιτρέψουν να πετύχουμε ευρία υποστήριξη για την έκθεση όταν θα ψηφίσουμε σε μία ώρα περίπου. Και νομίζω ότι αποτελεί καλή βάση για τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει με θετικό μάτι αυτό το έργο που επετελέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξ των Πρασίνων, το λόγο έχει για δυόμιση λεπτά η κυρία Τρουπέλ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλφιν για τη φιλόδοξη έκθεσή του και να σας επενθυμίσω για μία φορά ακόμα ότι το δικαστήριο ήταν εκείνο που είχε απαιτήσει η εξωτερική εντολή να καθοριστεί υπό συναπόφαση, δηλαδή έδωσε πιο πολλά δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ασφαλώς το καλωσορίζουμε ως ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δώσει πολλούς ε, καλούς στόχους στην στην συνθήκη της Λισαβόνα, καταπολέμηση της ένδυας, ε, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και το καθεξής. Είναι λοιπόν σωστό η ΕΤΕΠ ως μέσο ακριβώς να επιδιώξει τους σκοπούς αυτούς. Όχι να ταχθεί κατά αυτόν, αλλά να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο έχει προκειμένου να εφαρμοστούν οι στόχοι αυτοί, να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και μιλάμε κυρίως για περιβαλλοντικές υποδομές, για καλύτερη υπρευσή, για εγκαταστάσεις υγιεινής, για πιο πολλά μέσα, για την υγεία και την παιδεία, γιατί ξέρουμε ότι εκεί βρίσκεται η διασφάλιση του μέλλοντος των τρίτων χωρών. Και έτσι καταπολεμάμε και την ε, φτώχεια από πλευράς των πρασίνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το optional mandate, αυτό το, αυτή η εναλλακτική εντολή σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας και αν θέλουμε να πετύχουμε στην πολιτική μας κατά την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την ΕΤΕΠ. Και με χαροποιεί επίσης αυτό που πρότεινε ο κύριος Κάλφιν για την οικονομική ανακάμψη και την, ε, τον εκδημοκρατισμό στην Μεσόγειο, στην Τινησία και την Αίγυπτο ιδιαίτερα θα πρέπει να συνδράμει η ΕΤΕΠ και γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικές αυτές τις τροπολογίες τις οποίες θα υπερψηφίσουμε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μεγαλύτερη διαφάνεια στην ΕΤΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κάθε χρόνο θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Θέλουμε να υπάρχει πραγματική διαφάνεια. Θέλουμε πριν τη λήψη αποφάσεων οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλες ε, αντιταλμένες ε, οργανώσεις να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και θεωρούμε ότι αυτή η διαφάνεια θα συμβάλλει και στην αποδοχή της ΕΤΕΠ. Δεν πρόκειται να την υπονομεύσει και γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε με όλα αυτά τα καλά μέτρα τα οποία έχουμε προγραμματίσει το Συμβούλιο να υποστηρίξει αυτή την πολιτική προσέγγιση της ΕΤΕΠ. Ελπίζουμε να είναι γρήγορη η διαδικασία αυτή, η οποία θα αποβεί προς όφελος των πολιτών στις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ και τώρα ένα λεπτό. Η κυρία Σουίνμπερν από τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Εγγύηση για τέτοια δενοδότηση για προγράμματα εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχει οικονομικέ συνέπειε. Όταν φαίνεται ότι χρησιμοποιούμε καλά τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι πραγματικά γίνεται σωστή ανάλυση του κινδύνου και έλεγχο για να χειριζόμαστε αυτά τα δάνεια και να δούμε τι στο ζύγιο πετυχαίνουμε. Σαν βουλευτέ πρέπει να έχουμε επίγνωση των ε, κινδύνων για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και για τον προπολογισμό των κρατών μελών. Συστήματα ελέγχου και διαφάνεια θα είναι κρίσιμη σημασία να χρησιμοποιήσουμε ε, σωστά αυτό το μέσο. Το είδαμε και με τη χρηματοδοτική κρίση. Οι τράπεζε δεν ήξεραν πάντα ποιε ήταν οι ευθύνε του και τι είχαν αναλάβει. Θα πρέπει να μάθουμε από εκεί. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν επικρατούν τα αναγκαία επίπεδα δημοκρατικού ελέγχου. Θα πρέπει αυτοί που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χειρίζονται αυτά τα προϊόντα τα και παίρνουν τέτοιε σημαντικέ αποφάσει ότι έχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για να χειριστούν αυτά τα θέματα. Είναι χρήματα των φορολογουμένων, πρέπει να τα ξοδέψουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σουίνμπορν. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς για δυόμιση λεπτά ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, σήμερα συζητάμε Συγχρόνως ε, το ζήτημα μιας ε, περαιτέρω διευκρίνησης που θα πρέπει να χορηγηθεί στην ε, ΤΕΠ αλλά και της ανάγκης χρηματοδότησης. Θεωρώ λοιπόν όλη η διευκρίνηση της εντολής και η διεύρυνση αυτής πως αναφέρεται στην πρόταση είναι μια πολύ καλή ιδέα θα μας επιτρέψει και θα πρέπει και στην τράπεζα να πετύχει καλύτερα και ασφαλέστερα τους στόχους για να βοηθήσει αποτελεσματικότερα στην συνεργασία και την ανάπτυξη. Έχουμε δει πως ε, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλουν να εξαρτώνται απόλυτα από τις, ε, τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης ε, αξιολόγηση μάλλον πιστοποιητικής ικανότητα, τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σωστά. Εάν θέλουμε όμως ε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν επενδύουμε σε ζητήματα υγείας, καταπολέμηση τη ένδυα και σε στόχους χιλιετίας, χρειάζεται να πούμε ότι, κοιτάξτε, συζητάμε και εξετάζουμε τη σχέση που έχουμε με τους 20 αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μεταξύ άλλων όμως, όχι αποκλειστικά, παραδείγματο χάρη. Γιατί να είμαστε τόσο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τις εγγυήσει που πρέπει να χορηγούν οι φορολογούμενοι, αλλά ξεχνάμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν φρόντισε να ρυθμίσει τις ε, ιδιωτικές επενδυτικές τράπεζες διότι θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες τους ήταν κατά το μάλλον ήταν εγκληματικές. Και τώρα να αναφερθώ σε ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχουν δισταγμοί, επιφυλάξει ε, με τις οποίες συμφωνώ. Αφενός υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια, μια διεθνή πολιτική, αλλά εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν χρηματοδοτήσει τη ΕΤΕΠ σε χώρε ε, όπως η Λιβύη και όχι στην ε, Λευκορωσία. Βασιζόμενοι μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα. ο ίδιο ισχύουν και εδώ και εκεί. Και, και στις δύο χώρε. Τώρα, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέτω το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν ε, μπορεί να παραβλέπει τους ε, στόχους της ε, ελευθερίας και δημοκρατίας. Το λόγο τώρα έχει στην κυρία Σέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρησιμοποιεί δημόσια ε, κεφάλαια των εθνών της, της Ευρώπης για να δίνει δάνεια είτε ε, σε 74 χώρες. Όταν συγκρίνεται με άλλα διεθνή ιδρύματα που έχουν παρόμοιες αρμοδιότητες, η ΕΤΕΠ και η φήμη της δεν είναι μια φήμη διαφάνειας και η πολιτική δημοσίευση στο κοινό δεν είναι ε, ακόμα επαρκής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κοινό ακόμα δεν γνωρίζει πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά και η έκθεση αυτή απαιτεί ακριβώς δημοσίευση των ενδιάμεσων τραπεζών που χρησιμοποιούνται ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά εγγυητής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαίος φορολογούμενους. Σας, καλώ να καταψηφίσετε την έκθεση αυτή και να υποστηρίξετε τα συμφέροντα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Ολοκλώνεται ο γύρος αυτός των ε, ομιλιών με τον, ε, κυρία... με τον κύριο Χάρτον. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει ο σοσιαλιστής ε, κ. Κάλφιν. Ε, το ΕΛΚ δεν θέλει να υπάρχει τέτοια δραστηριότητα ο προϋπολογισμός της ΕΤΕΠ εγγυάται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το φορολογούμενο και συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως η Γάζα, η Λιβύα, το Τουρκμενιστάν, η Κούβα και είναι όλες αυτές χώρες οι οποίες δεν λάμπουν, ξέρετε, διά της δημοκρατικής τους αντιμετώπισης και τώρα θέλουμε να αυξήσουμε το ανώφλι αυτό της ΕΤΕΠ και θέλουμε να επενδύσουμε για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Μα στη Γάζα, μα στην Κούβα. Θα γίνουν αυτά. Αυτό είναι υλικό για να κάνουμε καινούργια ταινία για το Mr. Bean. Όχι πολιτικός στόχος. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να το καταψηφίσετε. Ευχαριστούμε κύριε Χάρτονγκ. Ο κύριος Μπίρμαν ε, σήκωσε τη γαλάζια κάρτα Δεχόσαστε την ερώτηση, κύριε Χάρτον. Τέις, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ ε, πιστώσεων και ε, επιδοτήσεων δεν καταλαβαίνει ο κ. Χάρτον ότι η Ευρώπη δεν είναι ενίσως απομονωμένη σε όλο τον κόσμο και ότι αν θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα στην ε, Ήπειρό μα πρέπει να επενδύσουμε και σε άλλες χώρες. Ε, αυτό σημαίνει ε, Δεν το υποστηρίζετε αυτό κύριε Χάρτον. Κύριε Χάρτον, θέλει να απαντήσετε. Πρόεδρε, κύριε Μπέρμαν, ξέρω ασφαλώς ότι η πολιτική έχει να κάνει με τις πολιτικές επιλογές και εμείς επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε με πολύ πιο σωστό τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων στην, ε, πιο πολύ στην εξωτερική πολιτική των κρατών μελών παρά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Χάρδον. Περνάμε τώρα στους ε, επόμενους αγορητές. Ε, καταρχήν έχουμε την κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα που έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του σε ό,τι αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων οικονομικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των μηνυμάτων που μπορεί να αποστέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου. Χρειάζεται λοιπόν να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες υπέρ των πληθυσμών και η Ευρώπη η οποία ε, δρά μέσω της ΕΤΕΠ μπορεί να προσφέρει σημαντική στήριξη σε αυτή την μεταβατική περίοδο για να βελτιώσει τις υποδομές αλλά και να βελτιώσει τις ε, επιχειρήσεις η έκθεση σημερινή προβλέπει μια αύξηση των ανωτάτων ύψου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα, για τα χρήματα τα οποία δαπανά εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα να προχωρήσει σε σημαντικά προγράμματα ε, και την σταθεροποίηση των περιεχών της Μεσογείου αλλά και χωρών που ε, προτίθεται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. κυρία Ματέρα παρατηρεί ο πρόεδρο. Οι διερμηνεί παρατηρούν ότι διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούν να σα ακολουθήσουν. Διαβάζετε λίγο πιο αργά, παρακαλώ. Έτσι η δουλειά του θα γίνει καλύτερη. Ζητώ συγγνώμη. Για να πετυχθούν, έλεγα, οι στόχοι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα πολύ ψηλό ποσοστό συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτική Δράση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει μια, εξέταση, μια κοινή διακυβέρνηση στις χώρες όπου δράει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επιθυμώ να ε, δημιουργηθεί μια πλατφόρμα προκειμένου να μελετηθεί από κοινού και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο πώς να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ένωσης με χρήματα οικονομικά μέσα και με καινοτόμες μεθόδους. Λυπάμαι που δημιούργησα πρόβλημα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Ματέρα. Ενάμιση λεπτό, η κυρία Ερτζόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ΕΤΕ είναι ένα θέμα που εξετάσαμε με τους διάφορους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντική η εγγύηση των πιστώσεων που χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι βασικό φορέα εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω η ΕΤΕ όσον αφορά τη δανειοδότηση και θα αυξηθεί ο ρόλο τη περαιτέρω. Υπό τι παρούσε διατάξει, κανένας κανένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο δεν μπορεί να ελέγξει την ε, ΕΤΕ. Θέλουμε να το βελτιώσουμε αυτό γιατί εμποδίζει περαιτέρω ανάπτυξη. Η εξωτερική δανειοδότηση πρέπει να προσεχθεί περισσότερο από ότι η δανειοδότηση εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για λόγους που αναφέρθηκαν, αλλά επίσης διότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε με τον ίδιο τρόπο τις ε, διάφορες συναλλαγές εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο αυτές εντός. Άρα χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία για εξωτερικά προγράμματα. Ταυτόχρονα τα εξωτερικά προγράμματα είναι στρατηγική σημασία. Και καμιά φορά εφαρμόζονται σε πολιτικά σταθείς περιοχές. Σαν μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας θέλω να πω ότι τα ενεργειακά προγράμματα είναι πολύ σημαντικά. Πάνω από 50% των δανείων αφορούν αυτά τα προγράμματα και χώρες της ε, ε, ανατολικής εταιρικής συνεργασίας που είναι ζωτικό το συμφέρον εκεί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι οι εισαγωγές φυσικού αερίου προς τις χώρες της Βαλτικής και Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης προέρχονται από τις ανατολικές γειτονικές μας χώρες. Άρα είναι πολύ σημαντικό η ΕΤΕ να εστιάσει προστάσει τη στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που συνδέονται με τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό. Συμφωνώ με τον εισηγητή και τον συγχαίρω μάλιστα για αυτό που έκανε. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε στενότερη συνεργασία της ΕΤΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης και αυτή η συνεργασία μπορεί να προσθέσει σε αξία. Ο κύριο Λάμστορφ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική ανάπτυξης ε, αποκτά νέε αρμοδιότητες. Μία αναφέρθηκε. Συνοχή συνεκτική συμπεριφορά όλων των μέσων, όλων των ε, θεσμικών οργάνων. Και η συνθήκη της Λισαβόνας επίσης προβλέπει μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, πιο πολύ διαφάνεια, κοινέ αποφάσεις, συναπόφαση για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά θα κάνουν πολύ καλό σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα της συζήτησης και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ε, αρμόδιων επιτροπών καθήλυνση του Κοινοβουλίου. Ένα αποτέλεσμα της διαφάνειας είναι ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε για τη Λευκορωσία να διαγραφεί από τη λίστα των χωρών εκείνων στις οποίες μπορεί η ΕΤΕΠ να δραστηριοποιείται χωρίς να γίνει πρώτερη συζήτηση στο Κοινοβούλιο αν ε, τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν απελευθερωθούν οι αντιφρανούντες, αν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, ε, συνδικαλισμού και το καθεξής. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά ε, για μια χώρα η οποία συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια αυτά προτού δραστηριοποιείται η ΕΤΕΠ στη χώρα αυτή και χαίρομαι που ακολούθησε αυτή την πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι και καλό το Συμβούλιο να μας υποστηρίξει. Χτες συζητήθηκε μεταξύ των μέσων τι μπορούμε να κάνουμε. Και η κάθε Άστον είπε ότι θα πρέπει να αυξηθεί το πλαφόν το ανώφλι για την ΕΤΕΠΕ. Το Κοινοβούλιο το, το επιθυμεί αυτό, γιατί θέλει καλύτερη συνεργασία με την Τινησία, την Αίγυπτο, την Αφρική εν γέννη και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας αντίδρασης και το Συμβούλιο λοιπόν καλείται ανάλογα να δράσει. Νομίζω ότι με τα μέσα εξωτερικής δράσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μέσα με προσανατολισμό εμπορικό, μπορούμε να πετύχουμε, για παράδειγμα, στην Αφρική. Γιατί άμα υπάρχει ανάκαμψη, άμα υπάρχει και δημοκρατισμός, θα είναι πιο λίγοι οι μετανάστες. Γι' αυτό θα ήθελα να πω στον συνάδελφο ότι τα επιχειρήματά σας είναι πραγματικά βραχυπρόθεσμα και πρωτόγωνα, αν θέλετε. Η κυρία Χάουταλα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακολουθεί πολύ καλούς στόχους, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της φτώχειας. Φυσικά, η δραστηριότητα της τράπεζας θα πρέπει να συνάδει και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρά τρόπο ανοιχτό και διαφανή η τράπεζα. Και σε αυτό το πνεύμα οι πράσινοι υπέβαλαν τις τροπολογίες υπαριθμών 6 και 7 οι οποίες αποσκοπούν στη δημοσίευση όλων των ε, χορηγήσεων και στη δημοσίευση των πληροφοριών για όλα τα έργα στο ευρωκοινό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει ασφαλώς όπως και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, δημοσιεύει και τα ε, έγγραφά της. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Τώρα ένα λεπτό κύριος Τσαρνέσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η ΕΤΕ είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί? διότι οι φορολογούμενοι συμβάλλουν στη διάθεση των πόρων που διαθέτει Γι' αυτό πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής η τράπεζα. Πρέπει η τράπεζα αυτή ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δείχνει ποια είναι η λειτουργία της, οι επιχειρήσεις της με κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ως εκπρόσωπος χώρας που γειτονεύει με τη Λευκορωσία ότι είμαι υπέρ παγώματος δανείων, δυνατότητας χορηγήσεως δανείων υποστήριξης για το καθεστώς του Λουκασέγκου. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά για μας παντού, είτε είναι στις ανατολικούς μας γείτονες, στην Αφρική, την Ασία. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ε, η συνάδελφος Μοργκάντη. Ο συνάδελφος Μοργκάντη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτή την έκθεση θέλουμε να δώσουμε κοινοτικέ εγγύσει για τη χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων τη ΕΤΕ. Πολλέ επενδύσει που υποστηρίζει η ΕΤΕ λαμβάνουν χώρα σε χώρε που αυτέ τι εβδομάδε βρίσκονται στο επίκεντρο των ε, πολύ σημαντικών αλλαγών όπου ανετράπησαν αυταρχικά καθεστώτα από λαϊκά κινήματα. Θέλουμε να, να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε και σε άλλε χώρε τι κοινοτικέ εγγύσει. Εκεί όμω που υπάρχει υπονοία όσον αφορά το πόσο δημοκρατικέ είναι. Θα ήταν παράδοξο να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και διερωτώ με μήπω θα ήταν πιο χρήσιμο η ΕΤΕ να αυξήσει τι επενδύσει τη στην Ευρώπη να επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση μικρομεσών επιχειρήσεων, παραδείγματο χάρη, όπω. Ο ίδιο ο Επίτροπο Ταγιάννη εξέφρασε αυτή την επιθυμία την περσμένη Δευτέρα στην Ολομέλεια. Κλείνοντα, δεν μπορώ παρά να σημειώσω με απογοήτευση συμπερίληψη τη Τουρκία ανάμεσα στι υποψήφιε χώρε για πονταξικέ διεργασίε. Εμεί, τη Λέγκα του Βορρά, δεν θα δεχθούμε ποτέ, και υπογραμμίζω, ποτέ, η αδίποτε υποχώρηση προ αυτή την κατεύθυνση επ' αυτού και άλλων μετόπων. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Για ένα λεπτό, ο κύριος Στογιάνοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε πως ε, η έκθεση αυτή έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να δαπανώνται και σπαταλώνται χρήματα των Ευρωπαίων ε, φορολογουμένων ακόμα και, για την... ακόμα και στην Τουρκία. Εγώ υποστηρίζω αυτό που είπε ο Λόρδος Ντάρμουτ. Πράγματι ένας ε, Βρετανός Λόρδος έχει μια κοινωνική συνείδηση πολύ πιο έντονη από ότι ο σοσιαλιστής Κάλφιν. Εμείς θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα των πολιτών μας, γι' αυτό έχουμε κλέγει. Και όταν θα έχουμε βρει λύση για τα προβλήματα των πολιτών μας, τότε θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε χώρες όπως Τουρκία και άλλες. Για 1,5 λεπτό, συγγνώμη, υπάρχει μια γαλάζια κάρτα. Κύριε Κάλφιν, θα έχετε την ευκαιρία να κλείσετε τη συζήτηση ως εισηγητής. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να προχωρήσουμε για να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω. Ο κ. Σταυράκα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή μα κύριο Κάλφιν για την εξαιρετική έκθεσή του. Δεν υπάρχει επιβολία κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι η σημερινή οικονομική κρίση ανέδειξε ακόμα περισσότερο το σημαντικό έργο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλο τη ΕΤΕΠ είναι επίση σημαντικό, αν και λιγότερο γνωστό, εκτός των συνόρων της ένωσης στην υποστήριξη των εξωτερικών δράσεων της ευρωπαϊκής ένωσης μέσω της εξωτερικής εντολής την οποία συζητάμε σήμερα. οι προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση πρώτον για αύξηση της διαφάνειας δεύτερον για εισαγωγή της ρήτρας ευελιξίας για πιθανή ανακατανομή των περιφερειακών πόρων τρίτον για ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ με την εξωτερική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης τέταρτον για επέκταση των επιλέξιμων χωρών και πέμπτον για αύξηση του ορίου χρηματοδότηση είναι προτάσει θετικέ πολύ χρήσιμε αναγκαίε και απαραίτητε. προτάσει με τι οποίε συμφωνώ και υποστηρίζω αγαπητοί συνάδελφοι γιατί και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του έργου τη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων αλλά και ταυτόχρονα βελτιώνουν τη θετική εικόνα και παρεμβατικότητα τη ίδια ευρωπαϊκή ένωση στον κόσμο. σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάν Μιούλτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν δεν μας ε, απατούν ε, οι ενδείξεις, ε, είναι όλο και πιο σημαντικός ο ρόλος της ΕΤΕΠ. Το σημαντικό για μένα είναι ότι ποτέ να μην τεθεί ε, ένα αμφιβόλο ή το τριπλό α με το οποίο αξιολογείται η Τράπεζα Επενδύσεων. Κοιτώντα τι συζητήσει για τι χρηματοπιστωτικέ προοπτικέ, ε, φαίνεται ότι η ποσότητα χρημάτων τα οποία, η οποία θα διατίθεται από τα κράτη-μέλη δεν θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που διατίθεται ήδη σήμερα και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να κοιτάξει πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά καλύτερα για να εκπληρώσει κάποιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το κάναμε και στο παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι εγγυήσει που δίνουμε στην ΕΤΕΠ και θεωρώ ότι θα είναι λοιπόν σημαντικό η τράπεζα το συντομότερο δυνατόν να υποβάλει μια σχετική έκθεση για να αναφέρει ότι κοιτάξτε αυτές είναι οι πιο επιτυχείς εγγυήσεις, παράγοντες πολλαπλασιασμού που έχουμε να καταδείξουμε. Έτσι μπορούμε και στις δημοσιονομικές προοπτικές να κοιτάξουμε και να επιλέξουμε ποια χρήματα θα επιλέξουμε και ποια project θα, επιτρέψουμε, θα επιλέξουμε για την ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ κύριε Μιλντερ. δεν ξέρετε, δεν μπήκε μπρο το χρονόμετρο, αλλά πιστό δεν έχει σημασία. Περαστικά είναι όλα αυτά. Λοιπόν, επόμενο αγορητή ο κ. Πορέμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε αισιόδοξοι όταν βλέπουμε ότι πρόσφατα η εξωτερική πολιτική ενισχύθηκε. Και τώρα έχουμε και νέα μέσα, όπως το προενταξιακό μέσο ή ε, το μέσο για την ε, γειτονία και τη συνεργασία. Η ΕΤΕΠ θα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία στις μεταφορικές υποδομές και τις ενεργειακές υποδομές, όπως ε, τον αγωγό Ναμπούκο και άλλους αγωγούς που είναι στατηγική σημασία. Η ανατολική εταιρική συνεργασία θα πρέπει να συνεπάγεται το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Λευκορωσία. Εάν η κυβέρνηση της Λευκορωσίας δεν στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι η σημαντικότερη υποχρέωση της κυβερνήσεως, τότε η χρηματοδότηση από την ΕΤΕ δεν θα πρέπει να χορηγηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ολοκλώσαμε αυτό τον γύρο και περνάμε τώρα στο γύρο του Catch the Eye. Έξι των αριθμών. Ο κύριος Σον Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πρόβλημα. Ας επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κυρίω όσον αφορά την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Σαν Ιρλανδό Ευρωβουλευτή, θεωρώ ότι είναι ηρωνικό ότι συζητάμε σήμερα το πρωί το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εγγυηθεί κατά των απολειών για έργα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βγάλει κέρδη από δάνεια που χορηγεί στην Ιρλανδία, σύμφωνα με το σύστημα υποστήριξης. Και το κέρδος είναι περίπου 3%, δηλαδή 5 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι κάτι βιώσιμο, δεν είναι δίκαιο και δεν νομίζω ότι είναι νόμιμο. Επίσης, βεβαίως, είναι απίστευτα δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς εμείς πρέπει να πληρώσουν 5,8% όταν δάνεια σε άλλες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήταν στα 3,2%. Με την νέα κυβέρνηση θα ζητήσουμε επαναδιαπραγμάτευση του θέματος. Και διακόπτω το μιλητή από τον Πρόεδρο. Ο κ. Πάσκα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότομη κύριε Επίτροπε, η διεύρυνση της εντολής ε, του ΕΤΕΠ, της ΕΤΕΠ ε, επιβεβαιώνει ότι η σημερινή ε, σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΤΕΠ αποδεδεί καρπούς σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την εντολή της ΕΤΕΠ. Επίσης, έχει να κάνει με τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις της ΕΤΕΠ που καλύπτουν τις δραστηριότητε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις δραστηριότητε, αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, αυστηρή μάλιστα. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιούνται για να επιτύχουν τους στόχους τους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας καλοκουρδισμένος και διαφανής μηχανισμός για την εποπτεία της επίτευξης των στόχων αυτών. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια για την χρήση των ε, στόχων. Ναι, λυπάμαι, λέει ο Πρόεδρος, τελείωσε ο χρόνος σας. Η κυρία... Ε, dziękuję panie przewodniczący. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά την άποψή μου, η δραστηριότητα της ΕΤΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις αξίες που είναι δεκτές στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την πολιτική γειτονία. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δεχτεί τη Λευκορωσία ως δικαιούχο χώρα των δανείων της ΕΤΕ. Αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δάνεια της ΕΤΕ, οι Λευκορώσοι θα πρέπει να σεβαστούν το κάτω δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι συνεπής όσον αφορά τη στάση της επ' αυτών. Θα πρέπει να επιβάλλει και οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντί έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα μέσο διακυβερνητικό τα κράτη-μέλη εγγυώνται και με τη σειρά της Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται για δραστηριότητε εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διατηρηθεί η αξιολόγηση 3α. Αυτή η εγγύηση είναι απόλυτα χρήσιμη. Θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέτοχος αυτής της τράπεζας για να μπορέσουμε να συγκεράσουμε το διακυβερνητικό με το κοινοτικό. Θα θέλαμε να δούμε το ύψος τώρα αυτός της ε, εγγύησης ε, ε, θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ και θα παρέχουμε και μια επιδότηση στην ΕΤΕΠ ανάλογα με τα προγράμματα που υποβάλλει. Και αυτή η εγγύηση, και τονίζω εδώ ότι η σχέση ανάμεσα στο Ταμείο Σταθερότητας τα 69 δισεκατομμύρια και τα 29, 29 δις νομίζουμε ότι φτάνουμε ήδη στο όριο των εγγύησεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοσλόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή αποτυπώνει πάρα πολύ καλά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διεύρυνση της εντολής για τις ε, εγγύησεις της ΕΤΕΠ είναι πάρα πολύ σημαντική και Ελπίζω ότι και η διαδικασία συνδιαλλαγής θα σταθεί με επιτυχία. Υποστηρίζω την ε, πρωτοβουλία για την ε, περιοχή της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη και όλα όσα συνέβησαν προσφάτως και συμβαίνουν ακόμη στην περιοχή και στη Λιβύη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την δημοκρατία στην περιοχή. Αφετέρου θεωρώ ότι η απόφαση να μην δοθούν εγγυήσεις και πιστώσεις προς τη Λευκορωσία είναι επίσης σωστή. Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά στη χώρα αυτή τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Κυρία Γκρέσλ, τελευταία ομιλήτρια. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε πριν εμπρός έναντι ενός νέου κύματος ε, εφαρμογής ε, σε ό,τι αφορά project της ΕΤΕΠ. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω. Ε, σήμερα 20 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός της ΕΤΕΠ και αν πληρούσαμε αυτά τα ποσά θα είχαμε προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν τα μελλοντικά χρήματα προς την ΕΤΕΠ να τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Δεν υπάρχουν Υπάρχουν 500 συνεργάτες ε, της ΕΤΕΠ ε, στο εξωτερικό, ενώ οι αντίστοιχοι συνεργάτες και υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάνω από 3.500. Θα ήταν πολύ καλύτερο να ελέγχονται τα συστήματα αυτά μέσω αυτών των υπαλλήλων. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσουμε να, πιστέψουμε, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση των κερδών και την δημοσιοποίηση των απολειών, των ζημιών. Θα πρέπει στις χώρες μας να εξηγήσουμε ε, και εδώ διακόπτει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Κάλλας ε, προκειμένου να απαντήσει στις διάφορες παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια σύντομα επιτρέψτε μου. Θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω τη σημασία του να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων βάσει της έκθεσης που κατά πάσα πιθανότητα θα υπερψηφιστεί σήμερα και θέλουμε να, έχει ληφθεί μια απόφαση πριν το καλοκαίρι για να μην βρεθούμε σε ε, μια φάση αναστολής των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το υπογραμμίζω εκ νέου. Επίσης, να σας διευκρινίσω, η ΕΤΕΠ δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες που έχουν καταστεί ιδιαίτερα σημαντικέ. Για παράδειγμα, η Αίγυπτος είναι μια χώρα που κατέχει μεγάλο ποσοστό των δραστηριοτήτων τη ΕΤΕΠ. 4,3 δις ευρώ της αναλογούν, κυρίως προς τον ιδιωτικό τομέα επίσης να διευκρινίσω κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες και ο προπολογισμό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μία τράπεζα ε, χρησιμοποιεί λεφτά των μετόχων. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά στην προκειμένη περίπτωση που καταβάλουν τα κεφάλαια και οι τράπεζες θα πρέπει να είναι υπεύθυνε και είναι υπεύθυνε για όλα τα χρήματα που έχουν δανείσει. Όλα αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν. Η κουλτούρα των τραπεζών αξιολογείται από τους οίκους αξιολόγησης και δύο φορές ακούσαμε σήμερα ότι η ΕΤΕΠ απολαμβάνει την πιο υψηλή αξιολόγηση και θα πρέπει φυσικά αυτό να επιδεινωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η κουλτούρα επαγγελματισμού. Είναι ένα σύμβολο των ευρωπαϊκών ε, οικονομικών. Θα πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει επίση έλεγχο. της ΕΤΕΠ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κρατημέλη συμμετέχουν στο σχετικό συμβούλιο. Μπορεί επίσης να περάσει από έλεγχο από τον Όλαφ και το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να γνωμοδοτήσει. Υπάρχουν λοιπόν ε, δημοκρατικοί μηχανισμοί για την άσκηση εποπτείας επί της τράπεζας. Επίσης να πω ότι η ευρωπαϊκή εγγύηση καλύπτει μόνο κάποιους πολιτικούς κινδύνους και ποτέ δεν έχει προκαλέσει απώλειες από το 1960 που δημιουργήθηκε για το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είναι λοιπόν ε, αξιόπιστο θεσμικό όργανο η ΕΤΕΠ. Φυσικά θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σε ποιους δανείζει και με τι κριτήρια δανείζει. Αυτά συζητάμε λοιπόν σήμερα και οι θέσει σας ασφαλώς ε, είναι απόλυτα σεβαστές και ασφαλώς και θα ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο εισηγητής Κύριος Κάλφιν, θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ΕΤΕ είναι θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ενώση, συμπεριλαμβάνεται στι συνθήκε Αβώνα ε, και ω θεσμικό όργανο θα πρέπει να βοηθά την επίτευξη των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε εντό είτε εκτό αυτή. Και εκείνοι που είπαν ότι η τράπεζα θα πρέπει να εμπλακεί σε ενέργειε εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι έχει εξωτερική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΤΕ ίσως να βοηθήσει την επίτευξη των αλόγων στόχων. Δεύτερον, η ΕΤΕ είναι χρηματοστικό ίδρυμα. Είναι πολύ σταθερό μάλιστα και όλες οι αλλαγές που έγιναν είχαν σαν στόχο τη διατήρηση σταθερότητά τη στις αγορές. Ταυτόχρονα δεν είναι αντίθετα αυτό με τη δυνατότητα ελέγχου και αξιολογήσεω των εξελίξεων των προγραμμάτων της ΕΤΕ και πώς επηρεάζουν το κλίμα. Δεν αυξάνει κάτι τέτοιο τον κίνδυνο, αλλά αντιθέτω τη διαφάνεια της τράπεζας. Σε αυτά που είπε Επίτροπος και που εκτιμώ τα όσα είπε, έχετε δίκιο κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι στο Συμβούλιο αναφέρθηκαν κάποια ευαίσθητα θέματα τα οποία συζητήθηκαν εκεί αλλά δεν αποφασίστηκαν. Πώς οι χορηγοί των τραπεζών και τα διάνοια Ευρωπαϊκή Ενώσης μπορούν να συνδυαστούν, πώ η Ευρωπαϊκή Αντεξιακή Βοήθεια μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη. Είναι ο μεγαλύτερο δωρητή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σαν ε, Ένωση, αλλά και σαν μεμονωμένα κράτη-μέλη και η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή. Δύο εναλλακτικέ έχουμε. Είτε να μην τα αντίξουμε το θέμα για την ευαίσθητο, ή να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε το Συμβούλιο για να βρούμε καλύτερη λύση και να αυξήσουμε την απόδοση όλων των πόρων που χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ την υποστήριξή σα και περιμένω ευρύτατη ε, συνένεση στο Κοινοβούλιο ε, και ότι θα περάσει το κείμενο αυτό μεγάλη υποστήριξη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ολοκλώθηκε το σημείο αυτό τη μισή διατάξεω. Θα ψηφιστεί σήμερα στι 12.00. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Προφορικέ ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.